Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Έχουμε προβλέψει ένα, μία ώρα χρόνο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Ε, δίωξη ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Κύριε Γκέρικε, έχετε το χρόνο. Κύριε Βάγγελ. Η προκάτοχό σα ε, η πρόεδρος, ε, έχασε μια ευκαιρία και δεν μου έδωσε δυστυχώς χρόνο Έτσι έχασε την ευκαιρία για μια πλήρως δημοκρατική συζήτηση. Είχα ζητήσει το λόγο στο Catch και δεν τον έλαβα. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε πιο δημοκρατικό διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Εναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια ε, του Προέδρου ή της Προέδρου της Συνόδου. Ο κύριος Γκέρικε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Μάιο του 2012 στο Μπακού είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision Light Your Fire κτλ. Ε, και όμως ήδη οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούσαν για έλλειμμα δημοκρατίας και ιδιαίτερα πλήττονται γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Και τις τελευταίες εβδομάδες ε, ακόμα και έμπειροι σχετικά με το Αζερβαϊτζάν έχουν συγκλονιστεί με τα όσα συμβαίνουν εδώ πέρα και τα οποία θα ήθελα να καταδικάσω. Αναμένω εγώ από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ξεκάθαρη φωνή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής γειτονίας και της οικονομικής μας πολιτικής. Η Άγκε Ένελκε, η Γερμανίδα παρουσιάστρια του, της Eurovision 2012, ήταν η μόνη η οποία είχε το θάρρος όταν ανακοίνωνε τους πόντους να ασκήσει κριτική στο Αζερβαϊτζάν. Και είπε επιλέξει καλές είναι οι εκλογές και το να δίνουμε πόντους ε, και καλή τύχη στο Αζερβαϊτζάν. Η Ευρώπη σας παρατηρεί. Και η Ευρώπη, θα ήθελα να πω στους Αζέρους, είναι και σήμερα στο πλευρό τους. Light your fire for human rights, που λέει και το τραγούδι. Ο κύριος Λάμσδορφ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι κυρία Πρόεδρε που σας βλέπω ε, και συγχαρητήρια και όλες ε, κύριε Επίτροπε για τον ε, διορισμό σας. Κυρίες και κύριοι είναι ανησυχητική η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ιράκ, είδαμε και άλλα μέρη, αλλά καλό είναι τώρα που στρεφόμαστε και σε αυτή την χώρα, όπου η κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς χειροτερεύει. Η κυβέρνηση ήδη έχει εντείνει την καταστολή στη χώρα αυτή, σύμφωνα με το Human Rights Watch και το Freedom House. Έχουν φυλακιστεί τουλάχιστον 40 πολιτικοί ακτιβιστές, περαστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και λοιποί με διάφορες επινοημένες ε, κατηγορίες, ε, φοροδιαφυγή, ναρκωτικά, ακόμα και προδοσία τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Ιούλιο που μας πέρασε συνελήφθησαν ε, οι σημαντικότεροι υπερασιστές ε, ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και πήγαν στη φυλακή μεταξύ των οποίων και ο κύριος, ε, η κυρία Γιονούς και ο σύζυγός της και ο Ιντιγκα Μαλίεφ ο σεβαστός επικεφαλής της, εταιρεία, της του ομίλου νομικής εκπαίδευσης και ποιο ήταν το έγκλημά τους έφτιαχναν έναν κατάλογο των ε, πολιτικών κρατουμένων και βρέθηκαν και οι ίδιοι στον ίδιο κατάλογο τελικά. Και υπάρχει επίσης ε, περαιτέρω περιορισμός της δραστηριότητας των ΜΚΟ. Πολλές ομάδες έκλεισαν αφού μπλοκάρισαν τραπεζική του λογαριασμοί. Από την άλλη, το Αζερβαϊτζάν καταβάλει κάθε προσπάθεια να αυξήσει το προφίλ του και σε μια κίνηση την οποία μπορώ να περιγράψω μόνο ως διαστροφική ανέλαβε την ε, προεδρία της ε, μιας επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και ο κύριος Αλίγεφ ήρθε και μας είπε πως όλα αυτά είναι ψέματα αλλά μετά από τέσσερις μήνες μόλις αποδείχθηκε πως είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει ο κύριος Βάιντεν Χόλτσαρ. Κοιτάξτε, το Αζερβαϊτζάν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτό είναι σημαντικό επίδομα για τη χώρα και για την Ευρώπη. Και βεβαίω ε, το βασικό κομμάτι του Συμβουλίου τη Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και εκεί πέρα πρέπει να μετρηθεί το Αζερβαϊτζάν. Παρά τι επίσημε διαβεβαιώσεις η κατάσταση επιδεινώνεται, περιορίζεται η δραστηριότητα των ΜΚΟ και οι άνθρωποι Αμάντο και καταδικάζονται. Ο κύριος ε, Φίλε όταν πήγε εκεί πριν από 15 μέρες είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι πρέπει να δούμε και αυτό το ψήφισμα. Μιλάμε για τις ε, περιπτώσεις ε, Αλίγευ και Γιουνούς και τις υπόλοιπες διώξεις. Πρέπει επίση να προειδοποιήσουμε το Αζερβαϊτζάν πω δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική αν συνεχιστεί η τωρινή πρακτική. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος να έχει το λόγο. Παρακαλώ να άψετε το μικρόφωνο. Μα αναμένο είναι. Δεν με ακούτε. Επαναλαμβάνω, ακούγομαι καλά. Ωραία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλή σας μέρα. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αναφίβολη δυστυχώς στο Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν είναι μία από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Μία χώρα πολύ σημαντική για τη γεφύρωση των σχέσεων με την περιοχή του Καυκάσου. Το γνωρίζουν αυτό οι συντάκτες του ψηφίσματος, ε, γι' αυτό και κατέληξαν σε ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο. Ε, αναφέρεται ιδιαίτερα η περίπτωση των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα, των πολιτικών κρατουμένων. Για παράδειγμα, ο δικηγόρος Ίντιγκαβ Άλιεφ, που είναι ε, υπερασπιστής και έχει υπερασπίσει πολλές υποθέσεις πολιτικών κρατουμένων, έχει υποστεί και ίδιο διώξεις. Πρόσφατα ε, στην Πράγα έλαβε το βραβείο Homo Hominae από τη μη κυβερνητική οργάνωση για τη People in Need. Σας να παρακαλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε το κοινό ψηφισμά. Σας ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τον, την άνοιξη του 2012 χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν ε, και διαδήλωσαν στον Πακού ζητώντας ειρηνευτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, αντίδραση κυβέρνηση ήταν ε, σκληρή καταπίεση με επιπτώσεις που τις βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Η κατάσταση κλιμακώνεται. Ε, δυστυχώς οι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές είναι θύματα αυτή τη δίωξη. Για παράδειγμα η Λέιλα Γιουνούς. Ενώ η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη προ την Ουκρανία και η δική μα προσοχή, η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν απολαμβάνει ατιμορρησία ενώ ε, αξιοποιεί του σιδηρογονάνθρακες που έχει. Έχουμε συμφωνία εταιρική σχέσης ε, ενώ διαπραγματευόμαστε συμφωνία σύνδεση με τη χώρα αυτή. Ποιο το νόημα αυτών των συμφωνιών αν δεν λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Αζερβαϊτζάν όχι μόνο δεν έχουμε καμία απόλυτο πρόοδο, αλλά έχουμε και παλινδρόμηση. Πήγε λοιπόν η διακοπή ε, των διαπραγματεύσεων, η αναστολή της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης και της εταιρικής σχέσης, ε, αν δεν υπάρξει πρόοδος. Αλλιώς όλα θα μείνουν επευτερώντα όλα τα ωραία λόγια που είπαμε. θα λέμε ότι θα διδράσουμε, ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Κοράω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν αυτή τη στιγμή έχει την εκπεριδριοπή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Όμως, το Αζερβαϊτζάν ε, παραβιάζονται συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα από την ελευθερία ε, έκφρασης, κυρίως στο διαδίκτυο και στην ελευθερία του συναθρίζεσαι. Ε, ο, το Αζερβαϊτζάν είναι ένα από του ε, ε, κύριους παρόχους φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Επομένω, ο στρατηγικό εταίρος μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν και τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον μα για τη δημοκρατική τους ε, υπόσταση και την διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από τι πιο σημαντικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που μα ενημερώνουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες ε, κρατούμενοι για λόγου συνείδησης επειδή εξέφρασαν την άποψή του, πρόκειται για δημοσιογράφους, blogger ή ακτιβιστέ Οκτώ κρατούμενοι ε, μεταξύ 18 και 30 ετών φαίνεται ότι κάνουν απεργία πείνα προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. Ζητάμε από την ε, Ευρώπη να πιέσει το Αζερβαϊτζάν ώστε να τηρήσει τα όσα έχει προσπογράψει στο, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Αζερβαϊτζάν είναι από τους πιο σημαντικούς ε, ε, εταίρους και λαμβάνει και πόρους για χρηματοδότηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, θα πρέπει να ζητήσουμε να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αλλιώς είναι σαν να καταδικάζουμε αυτά τα νέα παιδιά που κάνουν απεργία σπίνας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκοτ κάτω. Παρακολουθούμε με αποτροπιασμό ότι η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν διεξάγει πόλεμο κατά της κοινωνίας των πολιτών και κάποιων επιφανών υπερασιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ψευδοκατηγορίες. Αναφέρω την Λεϊλά Γιουνούς, το Αρίφ Γιουνούς, ε, Ρασέλ Γιασάροφ και Ινδιγά Μαλίεφ. Καταδικάζουμε την κράτηση των υπερασιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Αζερβαϊτζάν και είμαι υπερήφανη για το ότι οι πράσινοι πρότειναν ξανά την Λεϊλά Γιουνούς για το βραβείο Ζαχάροφ. Επίσης βλέπω πως η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια αποφάσισε να μην επισκεφθεί το Αφγανιστάν λόγω των πολλών εμποδίων στην ε, χώρα αυτή. Στο ψήφισμά μας ζητάμε να αποσυρθούν αυτές οι ψεύτικες κατηγορίες και ζητάμε επίσης να σταματήσουν οι επιλεκτικές ποινικέ διώξεις των επικριτών της κυβέρνησης. Επίσης ζητάμε να σταματήσουν ε, όλοι οι περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης ε, και του συνέρχεστε. Ζητάμε επίσης από την ύπατη εκπρόσωπο να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των ε, υπεραστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δοθεί περισσότερο βάρος στην κατάστασή τους. Επίσης επιμένουμε πως οι διαπραγματεύσεις ε, για μία στρατηγική εταιρική σχέση να παγώσουν μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία θέλουμε και να συνδεθεί η περαιτέρω σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ζερβαϊτζάν με τη βελτίωση των συνθήκων αυτών. Η περίπτωση Γιουνούς ε, μου επισημάνθηκε από μία ψηφοφόρο μου που την γνωρίζει και δεν πρέπει να την ε, ξεχάσουμε και πρέπει να μας ε, δώσει κίνητρο έτσι ώστε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του να εφαρμόσει αυτά τα οποία θα περιμέναμε και εμείς ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Δίνουμε τώρα το λόγο σε προσώπου των πολιτικών ομάδων, κυρία Τούν Ουντ Ευχαριστώ. Όσοι ερχόμαστε καθημερινά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης βλέπουμε την ε, ταμπέλα που μας δείχνει ότι το Αζερβαϊτζάν έχει την Προεδρία σε μια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε τις καταστροφικές ενέργειες ε, των αζερικών αρχών τους τελευταίους μήνες και παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν την παγκόσμια προσοχή που είναι στραμμένη προς την Ουκρανία για να καταπιέσουν τον δικό τους πληθυσμό το τελευταίους δύο μήνες. Πραγματικά έχει ε, φοβηθεί ο πληθυσμός, δεν τολμούν καν να κατεβούν στους δρόμους, δεν ε, ε, τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους κατά των πολιτικά, πολιτικών συλλήψεων. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, άμεσα να ενεργοποιηθεί ο ειδικό απεσταλμένος ε, και να κάνουμε και διαβήμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Επίσης με την αντιπροσωπεία μας στο Μπακού θα πρέπει να καταδικάσουμε απερίφραστα την κατάσταση αυτή και μάλιστα να απαγορεύσουμε την χορήγηση θεώρησης σε μερικούς υψηλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Αλίεφ. Θα πρέπει να επηρεάσουμε την κατάσταση του Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, ε, Δύο λόγια τι επιχειρήσει. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, αλλά δυστυχώ μερικέ από αυτέ ε, θα χρηματοδοτήσουν του πρώτου ευρωπαϊκά, τους πρώτους ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Μπακού. Γνωρίζουμε ότι έχει τεράστιο ρηκτό πλούτο, αλλά οι επιχειρήσεις αυτές ε, που πρόθυμα θα είναι χορηγοί έκαναν καμία έρευνα το κατά πόσο τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πραγματικά ο Αλίεφ έκανε μια προσπάθεια να παρουσιάσει υπό πολύ ρόδινο φω στη χώρα του, αλλά η κατάσταση δεν είναι έτσι στην πράξη. Και δύο λόγια ακόμη. Το ψήφισμα είναι πολύ καλό, αλλά είναι απλώ το πρώτο βήμα. Ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Πύρη. Er Σύμφωνα με την ε, Human Rights Watch τα τελευταία δύο χρόνια 40 υπραστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, blogger, δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί. Για αυτού τους ανθρώπους ζητάμε σεβασμό και την προσοχή μας βεβαίως. Είναι υποτίθεται στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη πολιτική γειτονία του Αζερβαϊτζάν. Όμω, υποτίθεται πώ η εταιρική μα αυτή σχέση βασίζεται σε κάποιε κοινέ αξίε τους προηγούμενους μήνες είχαμε ένα νέο κύμα σύλληψεων ανθρώπων που ασκούσαν κριτική στο καθεστώς. Αναφέρεται εδώ πέρα η Λέιλα Γιουνούς, ε, Ζαχάροφ και Αλίεφ. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, εφάρμοσαν τις αρχές ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ζητάμε από τις αρχές ε, στο ψήφισμά μας να απελευθερωθούν αμέσως οι πολιτικοί αυτή η κρατούμενη και να τερματίσει το κυνήγι μαγισσών ανθρώπων που απλά ζητά να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Τσαρνέτσκι. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα γίνετε πολύ καλή επίτροπος και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Βέβαια, θα χάσουμε εμείς ε, μια καλή Ευρωβουλευτή και Αντιπρόεδρο. Πάντως, ε, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή τύχη στις ακροάσεις. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση, γιατί ε, επικεντρώνει την προσοχή μας στις χώρες του Νοτιού Καυκάσου, που όπως είπαμε τον τελευταίο καιρό έχει διαφύγει της προσοχής μας, παρόλο που είναι πολύ σημαντική περιοχή. Και μιλώ ε, για τη σημασία που έχουν ε, οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις στις χώρες της, ε, του Νοτιού Καυκάσου. Εγώ πολύ συχνά έχω επαφές με εκπροσώπους της Γεωργίας, με Αζέρους και ε, σε πολλά θέματα έχουμε κοινέ απόψει και συμμεριζόμαστε κοινέ αξίε και αρχές. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη και ε, θα πρέπει ως ονόπο να έχουμε και συζήτηση για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, γιατί δυστυχώς σιωπούμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τσαρνέτσκι. Πολύ ευγενικά τα λόγια σας. Κυρία Κόνετσινα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα την χθεσινή ομιλία του κυρίου Σόλτς. Χρειάστηκαν 70 χρόνια στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την ιστορία της και το ιστορικό της παρελθόν. Το Αζερβαϊτζάν είναι ένα κυρίαρχο κράτος και προσπαθούμε να το αναγκάσουμε να ασπαστεί τις δικές μας αρχές περί δημοκρατίας. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας τέτοιας θέσης, γιατί το Αζερβαϊτζάν είναι κυρίαρχο κράτος και δικαιούται να αφιερώσει το χρόνο που χρειάζεται στη διερεύνηση και διαλεύκανση των υποθέσεων παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς όμως εξωτερική πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μια τέτοια στάση θα ήταν αντιπαραγωγική. Και επίσης αντιβαίνει στο πνεύμα συνεργασίας που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η αζερική κυβέρνηση είναι πολύ θαραλέα και θέλει να επιβάλλει κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Θα πρέπει να σεβαστούμε και το ιστορικό παρελθόν της χώρας αυτής ε, στο διάλογο που θα έχουμε. Πάντως είμαι πεπισμένη ότι η Επιτροπή της Βενετίας θα πρέπει να κρίνει κατά πόσο το Αζερβαϊτζάν τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε το Αζερβαϊτζάν να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις και όχι να οδηγηθεί στην καταστροφή. Ο κύριος Σέλη, ο κύριος Κέλλη, συγγνώμη, ο Κέλλη, όχι απουσιάζει, το λόγο έχει η κυρία Γκόμες. It's me? Yes. Okay. Please. Uh, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την απερίφραστη ε, καταδίκη ε, και στη λύτευση της αζερικής κυβέρνησης ε, που καταπιέζει όσους ε, δίνουν μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε χαλκευμένες κατηγορίες ε, και πολιτικά κίνητρα που χρησιμοποιούνται με απαράδεκτο τρόπο για να οδηγηθούν άνθρωποι στι φυλακέ με ψευδεί κατηγορίε κατοχή ναρκωτικών, κρυκτικών κτλ. Έχουμε επίση μία εκστρατεία εκφοβισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων και ακτιβιστών και Επίση, δεν λαμβάνονται υπόψη και παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει το Αζερβαϊτζάν να εφαρμόσει τι μεταρρυθμίσει που υποσχέθηκε ε, στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, στο οποίο είναι και μέλο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, την πολιτική εθελοτυφλίας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε ιδιαίτερες υποχρεώσεις ε, ε, και θα να απαιτήσουμε από το Αζερμπαϊτζάν να τηρήσει τις δημοκρατικές αρχές και να σταματήσει την κλιμάκωση της καταπίεσης. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση για τον εκδημοκρατισμό, αλλά αυτή η σχέση θα πρέπει να παγώσει σε περίπτωση που δεν δούμε θεαματικές πρόοδους από το Αζερβαϊτζάν θα πρέπει η αζερική κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσει πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε την διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι Δικαίω δίνουμε μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν και σε άλλε χώρε που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Ένας άνθρωπος, ένας ε, ε, εκπρόσωπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη φυλακή είναι ένας παραπάνω από όσο θα έπρεπε να βρίσκεται και θα πρέπει η συγκεκριμένη χώρα να σέβεται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφετέρου όμως θα ήθελα να τονίσω ότι το Αζερβαϊτζάν είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Η Ρωσία είναι δίπλα της, την πιέζει και το αυτό ισχύει και για το Ιράν. Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατηγικό εταίρο για μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, ιδίως ε, όταν πρόκειται για την ε, ε, κατοχή του Καραμπάχ και θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για το τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο, ο κύριος Μίμητσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν είναι όντω πολύ σημαντικέ και μάλιστα και στρατηγική σημασία σε ορισμένου τομεί. Βέβαια, μα φέρουν και ενώπιον πολλαπλών προκλήσεων. Έχουμε δύο κυρίω ανησυχίε. Γινόμαστε μάρτυρε σοβαρή επιδείνωση τη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Τους τελευταίους μήνες ε, πολλοί επιφανείς ε, προσπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήθησαν και φυλακίστηκαν μετά από συνεχείς ε, δράσεις καταπίσεις κατά της κοινωνία των πολιτών. Έχουμε επίσης κλιμάκωση και στην σύρεξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ και έτσι έσπασαν οι γέφυρες που δημιουργήθηκαν με την εκεχηρία του 1994. Φυσικά δεν μπορούμε να παραεκφράζουμε την ανησυχία μας για αυτές τις ε, ανησυχητικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, διαμάχη στον αγώνο Καραμπάχ. Ο Επίτροπος Φίλε και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ε, Σμιτ στην συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Αλίεφ και με εκπροσώπους των, της κοινωνίας των πολιτών στην πρόσφατη επίσκεψη στον Πακού συζήτησαν το θέμα της εταιρική σχέσης σε επίσημο υπουργικό διάλογο. Και τα θέματα αυτά ε, επισημάνθηκαν και από την, τον πρόεδρο Μπαρόζο που πήγε τον Ιούνιο στον Πακού. Και επειδή έχουμε ραγδαία επιδείνωση, έχουμε ενεργοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δώσαμε έντολες στο, στην αντιπροσωπεία μας να προσφέρει βοήθεια σε ακτιβιστές που υφίστανται κίνδυνο. Δυστυχώς ε, η καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών από το Αζερμπαϊτζάν αντιβαίνει στις ε, αρχές ε, της ανατολικής εταιρική σχέσης. Είναι σημαντικό να έχουμε μια θούσα κοινωνία των πολιτών για μια ευημερούσα δημοκρατία. Και επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους αζέρους εταίρους μας ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουν σταθερότητα και ευημερία της χώρας είναι μέσω ε, μιας ε, εύρυθμα λειτουργούσας ε, πολυκομματικής δημοκρατίας με ανοιχτή οικονομία και ανοιχτή κοινωνία. Φυσικά, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν με μια νέα νομικά δεσμευτική βάση και φυσικά θα πρέπει να εμπνευστούμε από κοινέ αρχές και αξίες και ιδιαίτερα από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης και εξυγχρονισμό της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, όχι μόνο στα πλαίσια του ρόλου του Αζερβαϊτζάν για την εξασφάλιση του ενεργειακού μας ανεφοδιασμού. Το Αζερβαϊτζάν λοιπόν που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, θα πρέπει να μεταρρυθμίσει την νομοθεσία και να λάβει υπόψη τις συστάσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών οργανώσεων προκειμένου η αζερική νομοθεσία να ευθυγραμμιστεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε ε, να μεταφέρουμε τα μηνύματα αυτά και φυσικά με συνεργάσιμο πνεύμα και εταιρικό. Και μετά από το, τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Γιάνγκλουν του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον πρόεδρο Αλίεφ, ε, προσβλέπουμε σε πρόοδο και σε επαφές και με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια του συνεδριάσου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δυστυχώς, η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχει συγκληθεί την τελευταία εξαίτια. Μια τέτοια συνάντηση θα ήταν ευκαιρία για επανάληψη του διαλόγου μεταξύ των αζερικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και η θέση εδώ σας περιμένει ο θόκος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μίμητσα. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος. Ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή και περνάμε στο επόμενο θέμα, το Μπουρούντι και ιδιαίτερα την περίπτωση του Πιέρ Κλαβέρ Μπονίμπα. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Μάρεκ Γιούρεκα, αλλά δεν το βλέπω στην αίθουσα. Ο κύριος Κοράου. Κοράου,